Meine Ο πρόεδρος Μπλοκ. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στην κοινή συνεδρίαση με την Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας. Έχουμε τη χαρά να συμπροεδρεύουμε με τη συνάδελφο Φώτιγκα. Θεωρώ ότι πρόκειται για σημαντικό θέμα γιατί βλέπουμε ότι αυτή η έλλειψη ασφάλειας που προκαλείται και με στρατιωτικά μέσα χρησιμοποιείται για την πρόκληση μεταλλαγών στις χώρες αυτές για να παρεμποδίσει κάποια λογική οικονομική εξέλιξη για την Ουκρανία. Αυτή η ανατροπή της ασφάλειας που προήλθε από την προσάρτηση της Κρυμαίας και από τις επιθέσεις στα ανατολικά της χώρας έχει επιτύχει το αποτέλεσμα να προκαλεί κόστος και ανασφάλεια ώστε να δυσχεραίνεται η αναγκαία πορεία μεταρρυθμίσεων της Ουκρανίας. Και με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ορισμένοι ότι επιτυγχάνουν τον στόχο ανατροπής των προσπαθειών μια θετικής εξέλιξης της Ουκρανίας. Βλέπουμε, είχα μάλιστα σήμερα την ευκαιρία να διεξαγάγω συζήτηση με εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης που εγκύπτουν στις θεσμικές εξελίξεις στην Ουκρανία. Είχα λοιπόν την ευκαιρία να συζητήσω πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει στήριξη του κρατικού μηχανισμού, να εξελιχθεί ένα σύστημα απονομής δικαιοσύνης που είναι σημαντικό για να λειτουργήσει και μια οικονομική εξέλιξη που θα οδηγήσει και σε μια βελτίωση των κοινωνικών συνθήκων. Αυτά οφείλουμε να τα δούμε και να δούμε ότι από πίσω κρύβονται ξεκάθαροι στρατηγικοί στόχοι. Η Γεωργία έχει αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα ήδη από το 2008. Πολιτική της Ρωσίας και απέναντι στην Απχαζία και την Νότια Οσετία. Και για τη Μολδαβία το ίδιο ισχύει για ακόμα περισσότερο χρονικό διάστημα, ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και την υπερδυνιστερία μέσα της οποίας γίνεται προσπάθεια άσκησης πιέσεων με επαναφορά συνοριακών θεμάτων ώστε να αναχαιτιστούν οποιασδήποτε οικονομικές προσπάθειες. Θεωρώ ότι βρίσκεται πίσω από όλα αυτά ένας αληθινός στρατηγικός σχεδιασμός και ότι οφείλουμε να συνδράμουμε τις χώρες αυτές και οικονομικά και τεχνικά για να μπορέσουμε να επιτύχουμε και την υποστήριξη των πολιτών. Η Ουκρανική κυβέρνηση έχει γίνει τώρα σάντουιτς ανάμεσα στις δυνάμεις κατοχής από τη μια μεριά και στους άλλους ανθρώπους από την άλλη μεριά προσπαθούν να προωθήσουν τις διαδικασίες μεταρρύθμισης και που απογοητεύονται γιατί δεν προχωρούν με αρκετή ταχύτητα. Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε σχετικά με το πώς μπορούμε να επιφέρουμε βελτιώσεις στην κατάσταση αυτή. Νομική μας βάση είναι η τελική πράξη του Ελσίνκη. Χαίρομαι που είναι παρόν ο Λαμπέρτο Σανιέ, Ζανιέ, πρόεδρος του ΟΑΣΕ, Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη. με τις προσπάθειες του οργανισμού από τη μια μεριά, αλλά και με την προσπάθεια που καταβάλει ο μηχανισμός που έχει προκύψει από τη Συμφωνία του Μίνσκ. Ο ΟΑΣΕ παίζει ρόλο κλειδί στα θέματα αυτά και σε ό,τι αφορά την νομική βάση και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της. εκφράζει τη χαρά μου που είναι παρόν και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Τζέιμι Σι, γιατί ο ΝΑΤΟ είναι σημαντικός φορέας τεχνογνωσίας για τα θέματα αυτά γιατί η συμφωνία του Μίνσκ παρόλες τις ατέλειές της αποτελεί τη βασική μας ελπίδα πρέπει να αντιληφθούμε και ποιος είναι ο στρατιωτικός σχεδιασμός της ε, Ρωσίας και να μπορέσουμε να οργανώσουμε την άμυνα των χωρών αυτών χωρίς βεβαίως σταθιωτική παρέμβαση του ΝΑΤΟ. Και Τζέιμι να σας πω ότι όλα αυτά τα γεγονότα, ιδίως στην Ουκρανία, έχουν οδηγήσει σε μια, πώς να πω, αναγέννηση του ΝΑΤΟ. Πράγματα τα οποία είχαμε ξεχάσει εδώ και 20 χρόνια, ότι δηλαδή χωρίς την Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία, τον ΝΑΤΟ, συλλογική άμυνα της Ευρωπαϊκής Υπήρου δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Χρειάζεται λοιπόν στενή συνεργασία και χαίρομαι, όπως είπα, που είναι παρόν ο GMC, αλλά και ο κ. Σέα από το Chatham House. Ο James Share. associate fellow του προγράμματος Ρωσίας και Βρασίας του Chatham House. Μήπως κυρία Φωτίγκα επιθυμείτε να τοποθετηθείτε. Α, θα θέλατε καλύτερα να λάβετε το λόγο στην, ε, στο πέραστο των συζητήσεων. Έχετε λοιπόν το λόγο κύριε Ζανιέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους συμπροέδρους Μπροκ και Φωτίγα θα αδράξω αυτή την ευκαιρία για να σας ενημερώσω για την κατάσταση σε πολλές περιφέρειες ε, του ΟΑΣΕ που απασχολούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια των συμφωνιών ε, ε, σύνδεσης και εταιρικών σχέσεων. Αυτό που βλέπουμε στις περιφέρειες και περιοχές αυτές μας βοηθά να δούμε με μία προοπτική της εξελίξης εδώ και 20 χρόνια. Από τις αρχές του, της δεκαετίας του 90 στον ΟΑΣΕ είχαμε πολλές ψυχρές παγωμένες σειράξεις που είδαμε μετά την διάλυση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που αποτελούσαν μία πρόκληση της νέας τάξης που είχε συσταθεί ως προς τα σύνορα, όπως διαμορφώνονταν, γιατί θα έπρεπε να διατρανώσουμε ε, ορισμένες αρχές του ΟΑΣΕ σε σχέση με την αεδαφική ακαιρεότητα και τα σύνορα των κρατών. Αυτά που είδαμε στην Αμπχαζία στη Νότια Οσετία, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και στην Υπερδνηστερία ήταν ότι υπήρχε μία, υπήρχαν ιδιαιτερότητες από τις εγχώριες σειράξεις, κάτι που σήμαινε ότι η διεθνής κοινότητα έπρεπε να καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να αντιμετωπίσει. Βλέποντας αναδρομικά τα πράγματα, έχουμε να κάνουμε με το γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλοι ε, διχασμοί και διαφορές στον ΟΑΣΕ και πολλές ε, διαφορές ως προς την οπτική μας γωνία και το πώς βλέπουμε τα πράγματα για τις ε, όλες διαδικασίες και το πώς αντιμετωπίζεται η ασφάλεια σε διάφορες πρωτεύουσες του ΟΑΣΕ. Αυτοί οι διχασμοί και διαφορές που βλέπουμε ανοιχτά και δραματικά στην Ουκρανία ήδη προϋπήρχαν σε προγενέστερη φάση σε σχέση με αυτές τις σειράξεις που προσπαθήσαμε να συγγίσουμε κάπως, να κατασυγίσουμε και να αντιμετωπίσουμε με συγκεκριμένους μηχανισμούς για να προσπαθήσουμε να δούμε τις ιδιαιτερότητες της κάθε κατάστασης. Η Ουκρανία έθεσε τα πάντα στα ίδια πλαίσια. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα προβλήματα έχουν παρόμοιες αιτίες. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε έχουν παρεμφερείς αιτίες. Βεβαίως η Ουκρανία μας το έθεσε αυτό κατά πιο δραματικό τρόπο το έφερε στο προσκήνιο, όπως είπε και ο Έλμαρ Μπροκ, σε σχέση με τις παραβιάσεις κανόνων, θεμελιώδεις κανόνες δηλαδή, που διέπουν τη σχέση των χωρών τα τελευταία 40 χρόνια. το θέμα της εγγύησης της εδαφικής ακεραιότητας, για παράδειγμα, είδαμε να καταρρύπτεται με την προσάρτηση της Κρυμαίας, παραβιάζοντας συγκεκριμένες εγγύσεις ασφάλειας που είχε δώσει προγενέστερα η Ρωσία στην Κρυμαία, στην Ουκρανία, πριν από την προσάρτηση βεβαίως της Κρυμαίας. Είδαμε λοιπόν ότι είχαμε να κάνουμε με μία καμπή, ένα σημείο καμπής σε σχέση με την σταθερότητα των κανόνων που διαπούν τις σχέσεις των ε, χωρών. Και η σύραξη στην Ανατολική Ουκρανία που αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα ε, εξαιτία της φύσης της είναι μια υβριδική σύραξη και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ορίσουμε τους πέκτες αν και έχουμε ενδείξεις για τους πρωταγωνιστές αυτή της εμπόλεμης σύραξης με βάση τις παρατηρήσεις και την επιτόπια παρουσία μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρόκειται για νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά περιπλέκονται περαιτέρω και οι διαδικασίες ε, επίλυσης των εμπόλεμων συγκρούσεων. Δηλαδή η Ρωσία και η Ουκρανία είναι δύο από τους facilitators της ε, φόρμουλας 5 συν 2 στην περίπτωση της υπερθμιστερίας Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό το πρότυπο έχει ε, πληγή κέρια. Και αυτό είναι μία λεπτομέρεια στην ε, όλη πολυσχηδή κατάσταση που αφορά την υπερθμιστερία όπου βλέπουμε ε, από τις πρόσφατες εκλογές στη Μολδαβία ότι φτάσαμε σε μια πιο περίπλοκη πολιτική εικόνα στην ίδια την ε, Μολδαβία. Σε σχέση δηλαδή με τις σχέσεις με την ίδια την υπερδνηστερία. Έκλεισαν τα σύνορα μεταξύ υπερδνηστερίας και Ουκρανίας και ε, Μολδαβίας και Ουκρανίας, ιδιαίτερα στον τομέα της υπερνηστερίας και αυτό οδήγησε σε αιτιάσεις από πλευράς υπερνηστερίας ότι προσπαθούν να, οι γείτονες χώρες να πνίξουν την οικονομία της χώρας. Αλλά αυτό ανεβάζει τις θερμοκρασίες σε αυτή την περιοχή και καθιστά τις συνθήκες πρόσφορες για μία οξύτερη φάση της ε, κρίσης και η όλη διαδικασία είναι πιο δύσκολη. Στην Απχαζία και την Νότια Οσετία είδαμε εξελίξει σε πολιτικό επίπεδο σε σχέση με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο αυτών περιοχών και της Ομοσπονδίας της Ρωσίας με μια σειρά ε, συμφωνιών που συνήφθησαν επίσης την οργάνωση των σχέσεων μεταξύ αυτών των περιφερειών και της Γεωργίας. Παρευρέθηκα στη Γεωργία πρόσφατα και ενώ εστιάζουμε την προσοχή μας στην κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και τους εξοπλισμούς που περνάνε από τη μία πλευρά στην άλλη, βλέπουμε πολλές φορές ότι οι εξοπλισμοί δεν ήταν στη ε, σωστή πλευρά των συνόρων και μιλώντας με έναν κάτοικο της ε, ε, Νότιας Οσετίας γεωργιανής προέλευσης μου έλεγε αυτό είναι το σπίτι μου και μου έδειξε πίσω αλλά μεταξύ αυτού και του σπιτιού του υπήρχε ένας φράκτης Σύμφωνα με τους αρχηγούς εδώ και τώρα, εάν θα πρέπει να ε, πάω να καλλιεργήσω τον αγρό μου, θα πρέπει να πάρω μια πτήση, ε, να πάω στην Τυφλίδα και μετά να γυρίσω πίσω στην άλλη πλευρά του Καυκάσου για να καλλιεργήσω το χωραφάκι, το μου. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ αποτελεί μια άλλη, ε, έναν άλλο τόπο σύραξης που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος επιτοπίως με εντατικοποίηση των διαφόρων συμβάντων. Δεν υπάρχει επαρκής δέσμευση των αρχηγών κρατών. Το ίδιο είδαμε και στην Αρμενία με οικονομικά ζητήματα, αλλά από πλευράς Αζερβαϊτζάν και ε, η, συμμετοχή, μάλλον η μετάβαση Αρμενίων στο Αζερβαϊτζάν δεν βοήθησε την κατάσταση, βοηθά την κατάσταση να επιληθεί. Άρα το περιβάλλον και εκεί είναι όλο ένα και πιο δύσκολο για την επίλυση διαφοράς. Τώρα, ως προς την Ουκρανία που είναι στο επίκεντρο των μελημάτων μας, δηλαδή είναι στο επίκεντρο των ε, προσπαθειών του ΟΑΣΕ. Συζητήσαμε τη διαδικασία του Μίνσκ πρόσφατα, ιδιαίτερα την πολιτική διαδικασία που είναι ύψη της σημασίας και πολύ δύσκολη, γιατί αν δούμε τις ε, προκλήσεις ε, με τις εκλογές αλλά και τη δυναμική του διαλόγου, βλέπουμε ότι είναι δύσκολο να το δούμε το όλο θέμα με τους αποσχιστές. Έχει αρχίσει όμως αυτή η διαδικασία διαλόγου, αυτό είναι το θετικό και συνεχίζεται. Υπάρχει δέσμευση, αλλά παράλληλα οι συζητήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες και παραμένουν δύσκολες. Ως διεθνής κοινότητα δεν μπορούμε παρά να διευκολύνουμε τη διαδικασία, δηλαδή να συζητηθούν αυτά γύρω από ένα τραπέζι, αλλά τα συμβαλόμενα μέρη είναι εκείνα που θα αποφασίσουν αυτά που απαιτούνται. Και θεωρούμε ότι έχουμε να διανύσουμε μεγάλη απόσταση ακόμα προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, τη στιγμή που η πολιτική διαδικασία ε, έχει εκινήσει, η επιτόπια κατάσταση μας ανησυχεί, γιατί φυσικά η ανακοχή κρατάει, καλά κρατεί υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν ε, μείζονες στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά υπάρχουν πολλές παραβιάσεις της ανακοχής ε, καθημερινά. Εκατοντάδες ε, παραβιάσεις ανακοχής και βλέπουμε ότι ολοένα και επεκτείνονται αυτές οι παραβιάσεις, αν και σε ορισμένες περιοχές έχει τη τελεστή πρόοδος, ιδιαίτερα στο νότο κοντά στη Μαριούπολη. Καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες έτσι ώστε να υπάρχει μία μεσολάβηση στην Ανατολική Ουκρανία για να φτάσουμε σε μία καλή διευθέτηση όπου ο ΑΣΕ θα είναι εγγυητής κατά κάποιο τρόπο ε, στην ε, ανακοχή στο Σιροκίνο και μπορούμε να το προωθήσουμε αυτό το σχήμα και σε άλλες πόλεις. Άρα μία πλευρά του ζητήματος είναι να παρέμβουμε για να μην υπάρχουν επιτόπιες σειράξεις και αν παγώσουμε την κατάσταση ε, φτάνουμε σε μία παγωμένη σύραξη η οποία δεν είναι κάτι το επιθυμητό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς έχει η πολιτική διαδικασία αυτή είναι μία προτεραιότητα και η ομάδα θεωρεί ότι το θέμα είναι ύψης της προτεραιότητας. Θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η πολιτική δέσμευση. Θα παραμείνω εδώ και μετά θα επεκταθούμε με τις ερωτήσεις των μελών. Ο πρόεδρος Μπροκ. Ευχαριστώ κύριε Σία. Κύριε Πρόεδρε, και βεβαίως και κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και πάλι που περιλάβατε το ΝΑΤΟ και το προσκαλέσατε στη σημαντική αυτή δημόσια ακρόαση. Χαίρομαι λοιπόν που επανέρχομαι εδώ. Μου δώσετε τώρα 10 λεπτά για να συζητήσω μαζί σας τρεις χώρες. Λίγο όπως το βιβλίο του Ιουλίου Βέρν σε 80 μέρες ταξίδι γύρω από τον κόσμο. Θα προσπαθήσω πάντως. Και πάλι όμως, παραλαμβάνω, είμαι μεγάλη τιμή για μένα να βρισκόμαι εδώ. Αντίθετα από την εποχή του ψυχρού πολέμου, η διαφορά σήμερα είναι ότι έχουμε έναν αριθμό χωρών ανάμεσα τη Ρωσία που φεύγει σιγά σιγά από την Δύση και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κοινότητες του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Τι γίνεται με τις χώρες αυτές? Μα αυτά δεν ρυθμίζουν μόνο την μοίρα τους, αλλά και τη μοίρα των μέλλον του ΝΑΤΟ, του Ευρωπαϊκού Project και το μέλλον της ίδιας της Ρωσίας. Όσο λιγότερο ασφαλής, τόσο πιο δύσκολα θα λειτουργούν οι χώρες αυτές. Και το εφέ της αποσταθεροποίησης θα είναι και στην περιοχή του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Ανεξαρτήτως τώρα των μελλοντικών προοπτικών ένταξης στο ΝΑΤΟ ε, την Ευρώπη των τριών χωρών που συζητούμε σήμερα, όσο πιο οικονομικά επιτυχημένες και πολυφωνικές θα είναι, τόσο περισσότερες πιθανότητες θα υπάρχουν ότι η Ρωσία θα εξελιχθεί και αυτή προς μια πιο φιλελεύθερη κατεύθυνση, έστω και πριν από την παρέτηση του Πούτιν το 2024. Τέλος πάντων την αποχώρηση καλύτερα του Πούτιν. Αυτό είναι βέβαια η κεντρική Ευρώπη. Υπάρχει αυτό το μήτελο Ευρώπα σήμερα και καταλαμβάνει και την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Δεν πρόκειται για ανταγωνισμό πλέον μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Το όραμα του ΝΑΤΟ που νομίζω το μοιράζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι οι χώρες μπορούν να έχουν πολλαπλές ιδιότητες. Βλέπετε την Τουρκία που είναι μέλος της Ανατολικής Συμμαχίας αλλά και της Ισλαμικής Ένωσης. Δεν είναι λοιπόν απαραίτητο να είναι ή το ένα ή το άλλο, είναι συμβατά τα πράγματα αυτά. Και η Ρωσία μπορεί να έχει στενές σχέσεις με τις χώρες αυτές, έχοντας ταυτόχρονα και στενές σχέσεις με τη Δύση. Αυτό δεν είναι ε, βεβαίως παιχνίδι μηδενικού αθρίσματος. Χώρες όπως η Γεωργία που έχει συμβάλει στο Αφγανιστάν και από τους μεγαλύτερους συνεισφορείς γενικά, όχι μόνο στο ΝΑΤΟ. Έχει συμμετάσχει σε κάθε μια από τις αποστολές του ΝΑΤΟ. Και η Ουκρανία ε, ε, προετοιμάζεται να παρέμβει μαζί μας στο Αφγανιστάν. Λοιπόν, αυτές οι εταιρικέ σχέσεις για να σημάνουν κάτι χρειάζονται και κάποια βοήθεια, κάποια αλληλεγγύη. Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια και να μην μείνουμε μόνο σε μια αντίληψη σφαιρών επιρροής και νέων γεωπολιτικών συμφωνιών όπου οι μεγάλες χώρες συνεργάζονται και οι μικρές υποχρεούνται να πάσχουν ό,τι αποφασίζουν οι άλλες. Ή αλλιώς θα αυξηθεί η όρεξη ορισμένων για γεωπολιτικές αλλαγές. Έχουμε λοιπόν πραγματικό γνήσιο συμφέρον να πράξουμε κάθε τι το δυνατόν για να στηρίξουμε τις χώρες αυτές. Ιδίω τώρα για την Ουκρανία, ο πρώτος στόχος πρέπει να είναι η σταθεροποίηση, όπως εξήγησε μόλις ο Γενικός Γραμματεύς Ζάνιερ. Είναι βαρύτατο το τίμημα 20% της οικονομίας της Ουκρανίας, 20% της οικονομικής της παραγωγής κατευθύνεται αλλού για την προμήθεια εξοπλισμών. Όπως είπε ο Ρομπέρτο, η κατάπαυση του πυρός και εκεί έχει παίξει ένα ρόλο ο ΑΣΕ κρατεί. Υπάρχουν όμως πολλά, πολλές απώλειες, έχουν 1.700 στρατιώτες νεκρούς, έχουν 900 ε, τραυματίες και έχουν μέχρι τώρα 560 παραβιάσεις της καταπαυσής του πυρός. Την ευθύνη φέρουν οι Ρώσοι. Όταν μιλούν οι Ρώσοι για, το, για τη συμφωνία του Μίνσκ, μιλούν σαν να είναι οι ίδιοι ουδέτεροι. Όχι, έχουν ευθύνη να φροντίσουν ώστε να λειτουργήσει η Συμφωνία του Μίνσκ. Πρέπει να αποχωρήσουν τα βαριά όπλα. Η Ουκρανία έχει κάνει θετικές προτάσεις για να απομακρυνθούν και όπλα μικρότερου διαμετρήματος, τα οποία οι αποσχιστές ακόμα δεν το έχουν συζητήσει. Έρχεται και η περίοδος του καλοκαιριού και ελπίζω να μην ξαναπάρει φωτιά η περιοχή. Στην περιοχή του Ντονέτσκ και αλλιού μόνο 10% των μαχητών, λένε οι Ουκρανοί, είναι ουκρανικής καταγωγής, είναι οι ντόπιοι. Οι υπόλοιποι 90 είναι ή Ρώσοι στρατιώτες ή πρόκειται από άλλες περιοχές. Άρα πρωτίστως απαιτείται επαγρύπνηση για τη Συμφωνία του Μίνσκ. Δεύτερο, ανεξαρτήτως των δυσχερών συνθήκων, πρέπει να προχωρήσει από η αποκέντρωση στην Ουκρανία. Να γίνουν τοπικές εκλογές υπό την ισχύ του Ουκρανικού Συντάγματος. Αυτό θα είναι το κλειδί για να ανακτηθεί ο έλεγχος στο ανατολικό μέρος της χώρας. Και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις τώρα, η Ουκρανία έχει κάνει πολλά πρόσφατα για να σπάσει τα μονοπόλια, για να αγωνιστεί κατά της διαφθοράς ορισμένων, ορισμένων ε, περιφερειακών κυβερνήσεων. Και κυρία και κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω την Ευρωπαϊκή Ένωση για την θαυμάσια δουλειά που έχει κάνει για να επιτρέψει να διαφοροποιηθούν οι πηγές για την Ουκρανία, οι πηγές ενέργειας δηλαδή για την Ουκρανία. Και βέβαια η Ουκρανία φιλελευθεροποιεί την ίδια της την αγορά. Μπορεί να παραγάγει και περισσότερο φυσικό αέριο, άρα θα χρειάζεται λιγότερο από αυτό που της προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τον ΝΑΤΟ κάνουμε και εμείς πολλά πράγματα. Έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα δημιουργίας αμυντικών ικανοτήτων. Στο Κίεβο επίσης εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε για μια εθνική στρατηγική, ένα στρατηγικό στρατηγικό δόγμα για να καταστήσουμε τις ε, Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, να τις φέρουμε δηλαδή σε επίπεδο του ΝΑΤΟ. Και άλλοι σύμμαχοι όπως Ενωμένο Βασίλειο, Ενωμένες Πολιτείες, Καναδάς, εκπαιδεύουν την εθνοφρουρά στην Ουκρανία και ενεργούς στρατιωτικούς. Και στην cyber defense, στην κυβερνοάμυνα, ενισχύουμε τις προσπάθειες με εκπαίδευση και με παρακολούθηση του εναέριου χώρου και στατιωτικού και μη στατιωτικού. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι η Ουκρανία, έστω με κάποια καθυστέρηση, να συνεχίσει την πορεία των μεταρρυθμίσεων. Αυτό είναι απόλυτα σαφές. Και οι ηγέτες της κυβέρνησης να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τρόπον που δεν έπραξαν οι παλαιότεροι ηγέτες του κράτους και της κυβερνήσεως. Να βοηθήσουν την Ουκρανία δηλαδή να επωφεληθεί από την ελευθερία που χαίρει μετά από τα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Για τη γεωργία τώρα. Στον τύπο. Αλλά και στον Washington Πόστ πιο πρόσφατα. Βλέπω άρθρα που λένε ότι οι Γεωργιανοί αρχίζουν και απογοητεύονται από την ένταξη της χώρας τους στους βορειοδατικούς θεσμούς που διαρκεί πολύ και θα χρειαστεί και άλλο χρόνο. Αρχίζουν και υποστηρίζουν λιγότερο λοιπόν τις εμπορικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχίζουν και υποστηρίζουν περισσότερο μια συμμετοχή στον ρωσικό ευρασιατικό χώρο. 31%. Και υπάρχει και η Eurasian Choice με 60.000 μέλη, σύνδεσμος δηλαδή πολιτικών σχηματισμών. και που ψάχνουν ένα είδος συμφωνίας με τη Ρωσία. Στη Μολδαβία βλέπουμε χωρισμό της κοινή νόμης περίπου στα μισά, 50-50, υπέρ ή κατά, αναλόγως της ε, ευρωπαϊκής πορείας της χώρας αυτής. Χρειάζεται να καταβάλουν προσπάθειες λοιπόν για να συνεχιστεί η διαδικασία, να συνεχιστεί η πορεία αυτή και να γίνει η μακρινή αυτή προοπτική μια γνήσια, αληθινή προοπτική, ιδίως στο παρόν περιβάλλον. Μιλήσατε ήδη για το ότι οι Ρώσοι χτίζουν φράχτες γύρω από την Οσετία. Πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς ότι δεν θα δεχτούμε οι οντότητες αυτές να εμφανιστούν ως κράτη. Όποιες ψευδοσυνθήκες και αν κάνουν, όσες ψευδοεκλογές και αν κάνουν εκεί. Πρέπει να μείνουμε σταθεροί για υπέρ της εδαφικής ακερότητας της γεωργίας. Δημιουργούμε και έξω από την τυφλίδα κέντρα εκπαιδεύσεως, κάνουμε και ασκήσεις και στην Μαύρη Θάλασσα και online με τις ε, γεωργιανές ενόπλες δυνάμεις. Η Γεωργία είναι ένας από τους πέντε special partners για ειδικέ δραστηριότητες, καθιστούμε σαφές δηλαδή ότι εργαζόμαστε έτσι ώστε και οι γεωργιανές ενόπλες δυνάμεις να αρθούν στο επίπεδο, στο ύψος μάλλον του επίπεδου των νατοικών δυνάμεων. Το ερώτημα θα είναι βέβαια τι κάνουμε στην επόμενη διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία για τη Γεωργία. Εν ώψη και της μελλοντικής πορείας ένταξης του Μαυροβουνίου. Για τη Μολδαβία τώρα, διαφορετική υπόθεση. 60 δευτερόλεπτα. Σας το υπόσχομαι. Μόνο 90% θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Και την πολιτική αυτή την υποστηρίζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Βέβαια, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ΝΑΤΟ, κατευθυνόμαστε πριν προς μια πλήρη ένταξη ο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωση κατά πάσα πιθανότητα από την άποψη αυτή θα είναι πιο σημαντικός. Ιδίω και εν ώψη των ε, συμφωνιών συνδέσεω με την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως η άρση των περιορισμών για την έκδοση προξενικών θεωρήσεων. Τώρα, η Μολδαβία βέβαια υφίσταται σημαντικές ρωσικές πιέσεις. Για παράδειγμα, για τους Κοκάσιους που υποστηρίζονται από τους Ρώσους και που η Ρωσία απειλεί ότι θα διώξει τους Μολαβούς που εργάζονται στη Ρωσία για να επιστρέψουν και το ίδιο με το θέμα της ενέργειας. Εκεί πρέπει επίσης να βοηθήσουμε με επιτόπου γραφεία συνδέσεως, με συνεργασία σε cyber defense κλπ. Πέντε πολύ σύντομα σχόλια τώρα για το μέλλον. Πρώτο, όσο κάνουμε περισσότερα στη βάση σεναρίων υβριδικών πολέμων και μιλούμε για ανθεκτικότητα, για κρίσιμες υποδομές, για στρατηγικές επικοινωνίες, ενέργεια κλπ. Πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο της ανθεκτικότητας και να μεταφέρουμε την εμπειρία μας αυτή και στους εταίρους μας που ίσως να τη χρειάζονται και περισσότερο από ότι εμείς οι ίδιοι. Δεύτερο, δημιουργία αμυντικών ικανοτήτων. Πρέπει να γίνει μια πραγματική επιτυχία. Δεν αρκεί να συμπληρώνουμε τετραγωνίδια. Να δούμε ποιες είναι οι πραγματικέ εκροές, το output. Χρειαζόμαστε καλύτερο συνδυασμό των μεμονωμένων προσπαθειών των συμμάχων και του ΝΑΤΟ. Τέταρτο, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργαστούν πιο στενά, ώστε να μην ακολουθούμε παράλληλε οδού αλλά να δημιουργήσουμε συνέργειε. Και τέλο να ενθαρρύνουμε τις χώρες αυτές να συνεργαστούν περισσότερο σε περιφερειακό επίπεδο. Όπως σε περιφερειακά πλαίσια στο παρελθόν, όπως το ΟΑΜ. Ζητώ συγγνώμη που κατανάλωσα κάπως περισσότερο χρόνο. Αλλά τα κατάφερα νομίζω και παράλληλα αυτά γρηγορότερα από ό,τι 80 ημέρες γύρω από τον κόσμο. Δεν μας είπες ακόμα ποιο είναι το, η λέξη στο Λονδίνο στην οποία συμμετέχεις. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε και κυρία Πρόεδρε, Χαίρομαι πολύ που έχω προσκληθεί και πάλι εδώ και παρευρίσκομαι και πάλι. Ω συνήθως ε, θα μιλήσω για τα θέματα αυτά κατά θεματικέ ενότητε. Τέσσερα σημεία θα ήθελα να θέσω. Το πρώτο σημείο είναι ότι και ε, στις τρεις χώρες ε, που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Μολδαβία, Ουκρανία και Γεωργία, η ηγεσία της Ρωσίας εξακολουθεί να ε, το βλέπει ότι είναι μια αντεπίθεση στρατηγική ενάντια στην ε, ε, δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πολλά χρόνια για να αποκλείσει τη Ρωσία από τον ιστορικό στρατηγικό της χώρο και να ε, υπονομεύσει, να αποσταθεροποιήσει το καθεστώς της Ρωσίας και το δικό της σύστημα αξιών. Για το ρόλο αυτό, το Κρεμλίνο θεωρεί ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία θεωρεί ότι δεν είναι από μόνο του πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι και κρίσιμο σε μια προσπάθεια να αλλάξει την τάξη ασφαλείας της Ευρώπης ε, επί τη βάση των αρχών της αποκατάστασης, ε, του συσχετισμού δυνάμεων και σεβασμού μεταξύ ε, μεγάλων και σημαντικών ισχυρών πόλων του διεθνού συστήματος. Ε, και δεν, βέβαια φυσικά θεωρεί ότι ε, τα συμφέροντα είναι πάρα πολύ σημαντικά και ότι είναι πιο σημαντικά από τους πολιτισμούς και από το αξιακό της ε, σύστημα. Ένα παράδειγμα είναι η αποκατάσταση του συστήματος της Γιάλτας. Κατά, τα, κατά τους τελευταίους μήνες ο ε, Ναρίσκιν που είναι ο ε, πρόεδρος της ε, Δούμα είπε ότι η επιλογή είναι ή θα ξαναμάθει ε, τα μάθημά της από τη Γιάλτα ή θα υπάρξει πόλεμος και ε, δεν ε, λέω ότι θα επιτύχει τους στόχους, τους, ε, τους στόχους της η Ρωσία, όμως είναι ρεαλιστικό και είναι ενδεχομένως και πιθανό ότι θα μπορέσει να, να, να, να, φτάσει σε μια κατάσταση, σε ένα αποτέλεσμα από το οποίο θα χάσουμε όλους. Έχει, διαχω, έχουμε, έχει διαχωρίσει τη θέση της η Ρωσία ως ε, τεράστιος εμπειρογνώμονας στο να ε, καταφέρνει μια κατάσταση στην οποία όλοι χάνουν ε, και αυτό που κάνει είναι να υπονομεύει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο ε, το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης αυτής, αλλά και εκεί που έχει συμβεί ήδη. Δεύτερο σημείο που θα ήθελα να θέσω, τα μέσα που χρησιμοποιούνται δεν είναι καινούρια, αλλά προσαρμόζονται βάσει των νέων συνθήκων και σε διαφορετικούς συνδυασμούς και με διαφορετικούς τρόπους που είναι τελείως καινούργιοι και αποσταθεροποιητικοί για μας και συμπεριλαμβάνουν ε, έναν ε, πόλεμο ε, πληροφοριών, τη διπλωματία, λόμπινγκ, πιέσεις σε διάφορα συστήματα συμμαχιών, τη χρήση του εμπορίου και της ενέργειας με καταναγκαστικό τρόπο, προβοκάτσια και εκφοβισμός ως στρατηγικό όπλο και όπως γνωρίζουμε τον αμφίσιμο ή μη γραμμικό πόλεμο, τον οποίο εμείς τον λέμε υβριδικό πόλεμο. Απλώς για να το επισημάνω, τι είναι υβριδικός πόλεμος πρώτη διάσταση να γίνονται κάπως πιο θολά τα όρια μεταξύ πολέμου και ειρήνης, ε, ε, θολά όρια μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών υποθέσεων και να προσπαθούμε να υπονομεύσουμε τους βασικούς πρωταγωνιστές ε, μία σύγκρουσης. Και όλα αυτά φάνηκαν με βάση αυτά που έγιναν στην Ουκρανία. Το «οι παγωμένες συγκρούσεις» είναι ένα σημείο που τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Τρίτο σημείο λοιπόν που θα ήθελα να θέσω. Οι συγκρούσεις αυτές ε, που τις έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ε, είναι ένα πυροτέχνημα, είναι μια νέα εφεύρεση της ε, ρωσικής πολιτικής, δεν είναι μια φυσική κατάσταση. Σε μερικές περιπτώσεις, για παράδειγμα στον Αγκόρνο Καραμπάχ, εκεί φαίνεται κυρίως αυτό, υπάρχουν λόγοι, υπάρχει γενή ε, αυτόχθονες, ε, υπάρχουν αυτόχθονες γηγενείς πολιτισμός που μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ε, ο λόγος αυτής της σύγκρουσης. Ένας άλλος τρόπος είναι η αποδυνάμωση της Μητροπολιτικής χώρας μέσω της καταστροφής της γειτονιάς ώστε να μπορεί η Ρωσία να είναι ένας ηγέτης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ε, σε διαπραγματεύσεις, ε, για πιέσεις ε, και ούτω καθεξής. Και όλες αυτές οι παγωμένες συγκρούσεις είναι ένα, ένας προάγγελος μερικών σποραδικών συγκρούσεων, όπως για παράδειγμα έγινε με την κρίση της Γεωργίας το 2008. Αυτός είναι ο στόχο τους, αυτή είναι η πρόθεσή τους. Ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες όλου αυτού του του, του, της προσπάθειας ε, ε, μεταφέρθηκε ε, στην Ουκρανία και είναι αναπληρωτής ε, ε, πρωθυπουργός στη λαϊκή δημοκρατία του Ντανιέσκο όπως την αποκαλούν λίγο μετά την κρίση της Ουκρανίας και μάλιστα πάρα πολλά ακραία στοιχεία λένε ότι η Ρωσία προσπαθεί να παγώσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, να τη σταματήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από μερικούς μήνες αποφάσισε ότι θα είναι επικοδομητική ότι θα αποδεχθεί την ρωσική πρόταση να μπει σε διαπραγματεύσεις σε σχέση με την μακροχρόνια εναρμόνιση της διαδικασίας, της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ευραφιατικής ολοκλήρωσης και θέλουν να κάνουν αυτή τη συζήτηση, συμφώνησαν ελπίζοντας ότι θα υπάρξουν δύο διεναρμόνισεις που θα μπορούσαν να συζητηθούν και ότι εμείς έτσι θα μπορούσαμε να διασκεδάσουμε τα άγχη της Ρωσίας. Όμως ο ρωσικός στόχος είναι εντελώς διαφορετικός. Τέτοιου είδους συζήτηση, κάθε είδους συζήτηση με αυτό το περιεχόμενο θα χρησιμοποιηθεί για να χρησιμοποιήσει, ε, να συνεχιστεί αυτή η παγωμένη σύγκρουση στη Μολδαβία, στην Ουκρανία και στη Γεωργία, ε, ώστε να υπάρξει μια ευρύτερη ε, συμφωνία η οποία θα μπορούσε να πάσα στιγμή ε, να καταρρεύσει γιατί θα είναι πλέον απίθανη. Και θα ήθελα να φτάσω στο τελευταίο, στο τελευταίο μου ε, σημείο. Δεδομένου λοιπόν ε, του πλαισίου αυτού, πώς πρέπει να αξιολογήσουμε την εξέλιξη της Συμφωνίας Μίνσκ 2 υπό το φως της Ουκρανικής κρίσης. Δεν θα σας πω τίποτε περίεργο αν σας πω ότι στο μεγαλύτερο τμήμα της Δύσης και σε επίσημο επίπεδο μάλιστα θα έλεγα υπάρχει μία εξίσωση ε, μεταξύ της σταθεροποίησης της σύγκρουσης στην Ουκρανία που είναι ένας στόχος ε, στον οποίο ο Τζέιμις μόλις αναφέρθηκε και ε, της συμφωνίας του Μίνσκ. Ε, και θα σας πω και κάτι που θα σας φανεί ενδεχομένως σε κάποιους από εσά αντιφατικό. Οι συμφωνίες ε, Μίνσκ δεν είναι μία βάση ε, σταθερότητας. Αυτό που κάνουν προσπαθούν να, θεσμο, θεσμοποιήσουν ένα, μια παγωμένη σύγκρουση με τους όρους που περιέγραψα προηγουμένως. Αν μελετήσει κανείς έχουν σχεδιαστεί από όσους τις ε, ε, διατύπωσαν και τις ε, διατύπωσαν στη Μόσχα πάρα πολύ προσεκτικά πριν κάποιες διατάξεις είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης ώστε να είναι εγγενώς ασταθής αυτή η συμφωνία και σας ε, διαβεβαιώ ότι είναι ασταθής. Μετά από όλες τις προσπάθειες της Ρωσίας στην Ανατολική Ουκρανία, οι αποσχιστικές δυνάμεις ε, συνεχίζουν να υφίστανται, ε, ελέγχουν όχι όμως πάνω από 5% της εδαφικής επικράτειας της Ουκρανίας, δεν είναι βιώσιμο αυτό. Δεν υπήρξε προσπάθεια της Ρωσίας να είναι βιώσιμη αυτή η κατάσταση. Τα ανθρωπιστικά οι ανθρωπιστικές ε, ε, ε, ομάδες έχουν καταφέρει να φτάσουν μεν, αλλά αν θεωρείτε ότι αυτή η κατάσταση θα παραμείνει και ότι θα, είναι, θα μπορέσει να γίνει βιώσιμη, δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει διοικητική αρμοδιότητα από όσους είναι επικεφαλής των περιοχών αυτών. Να τονίσω ότι η Ρωσία δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στις περιοχές αυτές ούτε και σε ολόκληρη την Ουκρανία και ότι η επίτευξη του στόχου που ανέφερε ο Τζέιμι Σί θα θεωρηθεί για τη Ρωσία μια στρατηγική ήττα. Και δεν υπάρχει καμία ε, σύγκριση, δεν υπάρχει καμία σύγκριση που να μπορεί να γίνει με την κατάσταση στη Γεωργία. Στη Γεωργία ε, η Γεωργία τα κατάφερε πάρα πολύ καλά με ε, την απόσχηση της Απχαζίας και της Νότιας Ουσουτίας και προσπάθησε να συγκεντρωθεί, ε, να συνασπιστεί γύρω από ένα μικρότερο, μια μικρότερη εδαφική επικράτεια για τους λόγους που ανέφερε ο Τζέιμι. Ο ε, υπάρχει δεν υπάρχουν εθνοτικές διαφορές ε, μεταξύ των ανθρώπων που ζουν στο Ντονιέσκ και μεταξύ εκείνων που ζουν στο Σλοβιένσκ. Ε, ε, η, Ανατολ... η Ανατολική Ουκρανία και η πιθανότητα, η υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν εκεί για την προσάρτησή τους από τη Ρωσία δεν είναι πάνω από 30%, διότι διαφορετικά θα είχε χαθεί ήδη η ε, Ουκρανία. Η Ρωσία λοιπόν έχει βρεθεί σε μια κατάσταση ε, που δεν τη θεωρεί ικανοποιητική είναι πολύ αποσταθεροποιητικό για ολόκληρη την Ουκρανία, κάτι το οποίο δημιουργεί τεράστια δυστυχία στους ανθρώπους εκεί, που δεν ικανοποιεί τους ε, υπέρ της απόσχησης ηγέτες ε, ούτε εκείνους, τους ικανοποιεί και βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία δεν ε, είναι μόνο πειρασμός, αλλά υπάρχει περίπτωση το πλεονέκτημα της εξουσίας να χρησιμοποιηθεί, να αξιοποιηθεί. Και ε, θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι εμείς πρέπει να περιμένουμε ε, εκπλήξεις και στην Ανατολική Ουκρανία και στην Ουκρανία στο σύνολό της. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να αρχίσουμε τη συζήτηση. Παρακαλώ εσείς κύριε Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ζήτησα το λόγο. Αλλά αφού με, μου ζητήσατε να πω λίγα λόγια, πρώτα να ευχαριστήσω τους παρεμβάντες. Είναι πάντοτε, πάντοτε εξαιρετικά ενδιαφέρον να ακούει κανείς τις διάφορες προσεγγίσεις οργανισμών όπως το ΝΑΤΟ ή ο Οργανισμός Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη και βεβαίως του εμπειρογνώμονος του Chatham House, τον οποίο γνωρίζουμε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας αυτές. Θα με ενδιέφερε ιδίως να ακούσω περισσότερα για τις παγωμένες συγκρούσεις. Είναι ενδιαφέροντα τα όσα είπε ο τελευταίος των παρεμβάντων για την συμφωνία του Μίνσκ μέσα στην οπτική αυτή των παγωμένων συγκρούσεων και, της, και την αντιμετώπιση που έχει η Ρωσία. Και θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις των δύο άλλων προσκεκλημένων για την σχέση, τον ορισμό ίσως, της ε, αξίας της συμφωνίας του Μίνσκ σε ό,τι αφορά τη διαχείριση μιας παγωμένης συγκρούσεως. Όντως έχουμε ανάγκη ενός ξεκάθαρου ορισμού μιας οριοθέτησης του προβλήματος και βρήκα πραγματικά ενδιαφέρουσα την τελευταία παρέμβαση που μας θέτει ενώπιον μιας ευαίσθητης καταστάσεως που έχει και διαστάσεις στρατηγικές σε ό,τι αφορά δηλαδή την κατάσταση όπως αυτή εξελίσσεται στα ανατολικά της, στο ανατολικό μέρος δηλαδή της Ουκρανίας. Επιθυμείτε να λάβετε το λόγο. Ε, ρωτώ γιατί την πρώτη φορά δεν είχε ζητήσει ο συνάδελφος. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Απευθύνομαι στον πρέσβη κύριο Ζάνιερ. Ευχαριστώ που είστε παρόν σήμερα εδώ. Βεβαίω και ανησυχώ για τα όσα συμβαίνουν στη γειτονιά της Ευρώπης. Και ιδίω με ενδιαφέρει όμως η εσωτερική ασφάλεια στην Ευρώπη. Και τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα εξτρεμιστικά στοιχεία. Μια από τις ρίζες είναι η Ισλαμοφοβία την οποία εκμεταλλεύονται ομάδες όπως Αλκάιδα και Ισλαμικό κράτος. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως Ευρωβουλευτές για να σας υποστηρίξουμε στις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλετε για την αποδυνάμωση αυτών των απειλών. Ευχαριστώ. Τάνοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε με ενδιαφέρον άκουσα τα περί νέου ρωσικού στρατηγικού δόγματος. Κάποια στιγμή ο Πούτιν είχε πει ότι θέλει να γυρίσει πίσω το ρολόι της ιστορίας και να επανακαθορίσει τις σφαίρες επιρροές στη βάση του μοντέλου της Γιάλτας. Και υπάρχει και ο κίνδυνος να κατεβάσει το κατόφλι χρήσης του πυρηνικού όπλου. Είναι ενδιαφέροντα τα όσα είπαν οι παρεμβαίνοντες ότι το μόνο που συνδέει Ρωσία, Κίνα, Ινδία και την Δύση είναι ο κοινό εχθρός των ακραίων μορφών τζιχαντισμού. Που απορροφά βέβαια για κάποιους τζιχαντιστές τα πολεμικά πεδία της Συρίας από τον Κάφκασο. Δεν ξέρω αν έμεινε σωστά τα τελευταία σχόλια του κ. Σέρ σε ό,τι αφορά τον ευνηδιασμό. Θεωρείτε ότι οι Ρώσοι θα κινηθούν γύρω από την Μαριούπολη για να προχωρήσουν προς τις μας. Η ερώτησή μου έχει βέβαια και μια ευρύτερη έννοια και απευθύνουμε στους κυρίους Σέρ και Σέι. Αυτή η προσέγγιση Ρωσίας και Κίνας και τα βλέπουμε αυτά ιδίω στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και εν μέρει και με την Ινδία μέσω του BRICS και της νέας τράπεζας BRICS και της, ε, του Οργανισμού Συνεργασίας της Αγκάης. Είναι πράγματι τρόπος αυτός αναζήτηση νέων συμμαχιών από πλευρά της Ρωσίας και θα είναι σταθερές οι σχέσεις αυτές δεδομένης και της εχθρότητας με χώρες όπως η Κίνα. Βλέπω και μια μαζική εκστρατεία με email κατά της συμφωνίας TTIP καθώς και χρηματοδότηση ακροδεξιών κομμάτων και ακόμη και αυτών των εκπροσώπων τους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την πλευρά εκείνη. Θέλετε να μιλήσετε από, την, ε, από τους φιλελευθέρους. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν ε, τόσα ε, ζητήματα που μπορεί να επηρεάσει η Ευρώπη για να επιλύσει τις παγωμένες σειράξεις. Με, ήδη με τις πέντε χώρες εταίρους στον ανατολικό χώρο, αλλά ίσως θα πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα των ελευθέρων θεωρήσεων, ιδιαίτερα με τη Μολδαβία. Αναφερθήκατε σε αυτό, γιατί μιλάμε για 75.000 κατοίκους της υπερθνιστερίας που τώρα έχουν διαβατήρια της Μολδαβίας και αυτό έχει επιπτώσεις και στην κοινωνία της υπερδυστερίας. Συμφωνείτε λοιπόν ότι το θέμα της ε, απελευθέρωσης, ε, της ελευθερίας ως προς τις θεωρίες θα μπορούσε να επεκταθεί στην Απχαζία, στην Νότια Οσετία και στην Ουκρανία. Και υπ' αυτή την έννοια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να θεωρήσει το θέμα της ελευθερίας των, ως προς θεωρήσεις ως ε, ένα τεχνικό καθαρά ζήτημα. Θα μπορούσε να έχει θετικές επιπτώσεις και για τις παγωμένες σειράξεις. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Εδώ και μερικά χρόνια στη Γεωργία δεν υπάρχει παρουσία του ΟΑΣΕ. Μπορεί να αποκατασταθεί η αποστολή για την Απχαζία και την Νότια Οσετή και ο ΑΣΕ μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην στερία. Γκάλερ. Ευχαριστώ. Περιμένω να φορέσετε τα ακουστικά σας. Νομίζω ότι οφείλουμε με λύπη να διαπιστώσουμε ότι η Ρωσία δεν τα καταφέρνει να διεξαγάγει μια πολιτική, να ασκήσει μια πολιτική που θα ήταν ελκυστική, ενδιαφέρουσα συναρπαστική για να προσελκύσει εταίρους να συνεργαστούν μαζί της. Προφανώς δεν μπορεί να το πράξει αυτό και επομένως καταφεύγει σε απειλές και αποσταθεροποίηση. Πρόκειται για πραγματικό γεγονός, το οποίο οφείλουμε δυστυχώς να διαπιστώσουμε παρόλη την ευρεία συνεργασία ή πάντως ευρύτατες προσφορές συνεργασίας που έχουν προέρχει από μας. Βρίσκω ότι αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Το ερώτημα τώρα είναι, πράγματι, τι κάνουμε στους διάφορους φορείς στους οποίους συμμετέχουμε, οργανισμούς που ασκούν πολιτική ή που διατυπώνουν προτάσεις πολιτικής. Διαπιστώνω ότι παραμείναμε ενωμένοι στην επιβολή κυρώσεων ως Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πλαίσιο βέβαια του ΝΑΤΟ έχουμε λάβει αποφάσεις που ελπίζω ότι μας καθιστούν ισχυρότερους και αξιοπιστότερους προς τα έξω. Και που στην αιχμή του δόρατος που έχουμε φτιάξει τώρα θεωρώ ότι αυτή είναι σημαντική για την αξιοπιστία. Τώρα πιο συγκεκριμένα για την Ουκρανία. Απευθύνομαι στον κύριο Ζανιέ και ρωτώ πότε θα έχουμε το αυξημένο αριθμητικά επίπεδο προσωπικού επιτόπου και τι μπορούμε να πράξουμε ώστε τα πρόσωπα αυτά να μπορούν να μεταβαίνουν ελεύθερα όπου επιθυμούν. Μεταξύ Τσιρόκινε και ρωσικού, ρωσικών συνόρων που είναι no-go area. Δεν μας αφήνουν να παίρνουμε εκεί. Τι δυνατότητες έχουμε να επιβάλλουμε την υποχρέωση αυτή στη Ρωσία που είναι μέλος του ΟΑΣΕ. Θα ήθελα επίσης να μας δώσετε μια εκτίμηση εάν είναι δυνατό να στεθεροποιηθεί η Ουκρανία με δική μας συμβολή ως χώρα με την έννοια ότι επιμένουμε στο status quo να σταθεροποιηθεί δηλαδή η γραμμή διαχωρισμού χωρίς να παράσχουμε οπλισμό στην Ουκρανία. Μπορεί να αντέξει η Ουκρανία πιο μακροπρόθεσμα να διατηρήσει στρατιωτικά το status quo. Ποια εκτίμηση έχετε. Αυτές είναι οι μου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων προς τους ε, τρεις ομιλητές για γιατί μετά τις ομιλίες τους δεν μπορούμε να είμαστε ούτε ουτοπικοί, ούτε να τρέφουμε αυταπάτες για την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης στρατηγικής πρόκλησης. Γιατί ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωσης και ΝΑΤΟ είναι το κλειδί για οποιασδήποτε μελλοντικές θετικές εξελίξεις για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη αστάθεια. Θα ήθελα αρχικά να πω, σύμφωνα με την παρουσίασή σας, ότι πρόκειται για μια προγραμματισμένη στρατηγική της Ρωσίας που εφαρμόζεται στις παγωμένες σειράξεις. Στην αρχή ήταν διεθνοτικές, μετά παγωμένες, μετά ξανανοίγουν όπως στην περίπτωση της Απχαζίας και της Νότιας Οσετίας και η de facto, ο de facto έλεγχος της Ρωσίας στην Απχαζία ε, Νότια Οσετία και η Περνιστερία με 160.000 στρατιώτες, στρατιωτικές δυνάμεις που μπορούν να φτάσουν μέσα σε δύο ώρες στο Κισινάου και ο έλεγχος των παγωμένων σειράξεων όπως ε, με τις ε, εταιρικές συμφωνίες που έχουν υπογράψει με την ε, επωνομαζόμενη αυτόνομη δημοκρατία της Νότιας Οσετίας και της Απχαζίας όλα αυτά δείχνουν ότι το ίδιο σενάριο ίσως ισχύσει και στην Ανατολική Ουκρανία. Προς τον κύριο Σύ είναι αυτή η ερώτηση. Κύριε Σύ, πώς ε, αντιμετωπίζετε την κατάσταση στην Κρυμαία που δεν είναι μια παγωμένη σύραξη, απλώς υπάρχει κατοχή, εδαφική κατοχή που έχει προωθήσει η Ρωσία. Πώς μπορεί να περάσει η Ρωσία από τη Μαριούπελη Μαριούπολη στην υπευνηστερία για να συμφωνήσω με τον κύριο Τάνοκ. Θα θέλαμε και τις ομιλίες σας γραπτός γιατί μας βοηθάνε πάρα πολύ για να είναι αντίβαρο στη μεγάλη ε, φιλορωσική παρουσία που υπάρχει και εδώ σε αυτό το σώμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε κύριε Μποστινάρο. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι παρουσιάσεις δεν ήταν ad hoc παρουσιάσεις. Αλλά θα το δούμε. Θα ζητήσουμε από τους ομιλητές ε, να μας υποβάλουν μένα γραπτά σχόλια εάν συμφωνούν. Ο κύριος Οστρεβίτσιους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σε όλους τους πανελίστ που βρέθηκαν εδώ και πρόθυσαν μία εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία. Στις εισηγήσει τους και θα ήταν σκόπιμο να διαδώσουμε αυτές τις πληροφορίες. Εξαιρετική η εργασία σας. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά την παρουσίαση του κυρίου Τζέιμι Σι. Είπε ότι η Ρωσία συμμετέχει άμεσα και θα πρέπει να λογοδοτήσει για τα γεγονότα της ε, Ουκρανίας. Όμως συμμετέχει και ε, στον ΟΑΣΕ και μαθαίνουμε για έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ ΟΑΣΕ και στρατιωτικών δυνάμεων της Ουκρανίας που βρίσκονται στην εμπροστοφυλακή μετά τους ελέγχους του ΟΑΣΕ επιτοπίως. Φαίνεται ότι πρόκειται για μία διαλκυστίνδα μεταξύ αυτών των θέσεων. Πώς θα μπορούσατε να σχολιάσετε τις κατηγορίες αυτές από πλευράς Ουκρανίας, γνωρίζοντας ότι η Ρωσία είναι παρούσα, παρέχει όπλα και υποστηρίζει πολιτικά τις κατοχικές δυνάμεις και δράσεις στην Ανατολική Ουκρανία. Δεύτερον, μία ερώτηση προς όλους τους ε, πανελίστ. Η Ρωσία δεν θέλει κανένα γείτονα που προχωρά σε μεταρρυθμίσεις. Είναι ιδιαίτερα ευτυχής με τις, ε, με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας γιατί δεν υπάρχουν μεταρρυθμίσεις σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Δεν έχουν προχωρήσει αυτές οι χώρες και έχουν τις ίδιες πολιτικές και κοινωνικές δομές, αν όχι χειρότερες, με 20 χρόνια πριν. Οι χώρες λοιπόν αυτές που θεωρούνται προευρωπαϊκές ή έχουν καλύτερες ε, δοκιμασμένες πρακτικές που είναι λειτουργικές, οι χώρες αυτές ε, δεν είναι αρεστές στη Ρωσία. Γι' αυτό με, τις παγωμένες, με μια παγωμένη σύραξη η Ρωσία τι κάνει στην ουσία προσπαθεί να αποσπάσει αυτές τις χώρες από τις μεταρρυθμίσεις. Ποια είναι τα μέσα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, όχι μόνο με ανθρωπιστική βοήθεια και αποστολές, καθώς και παρατηρητήρια. Πώς μπορούμε έμπρακτα να βοηθήσουμε με μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, έτσι ώστε να έχουμε μία προενεργή πολιτική. Γιατί δεν βλέπω μία φυλακή από τη δική μας πλευρά. Ο κύριος Φρονζουλίτσα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αν δούμε τη, λεκάνη του ευξήνου πόντου, βλέπουμε παλαιότερες παγωμένες συγκρούσεις ε, και νεότερες συγκρούσεις ε, με την Κρυμαία, για παράδειγμα, γύρω από τον ευξήνο πόντο. Φαίνεται ότι παίζουμε το παιχνίδι αυτό στην πλάτη του ευξήνου πόντου. Ε, ξέρουμε ότι η σημασία του ευξήνου πόντου ε, για την ευρακλαντική ε, σταθερότητα έχει αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Πρέπει να επικεντρώσουμε στην περιοχή αυτή τις προσπάθειές μας. Παράλληλα θα έλεγα ότι αν η Ουκρανία και η Γεωργία το 2008 ελάμβαναν την ιδιότητα μέλους τους στη Βουδαπέστη το 2008, ε, την, την ιδιότητα μέλους προς ένταξη. Θα ήταν διαφορετικά ίσως τα πράγματα. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε με διαφορετικούς τρόπους στη Ρουσία με στρατιωτικό, σε στρατιωτικό επίπεδο, με διάφορες κυρώσεις, οικονομικού χαρακτήρα, ε, προσπαθούμε τέλος πάντων να αντιμετωπίσουμε αυτήν την μεγάλη ασύμετρη και υβριδική απειλή που προέρχεται από τη Ρωσία. Αλλά θα ήθελα να επανέλθω σε ένα θέμα παλαιότερο, το οποίο είναι και πάλι σημαντικό. Πρέπει να απαντάμε στη Ρωσία με ένα σωστό τρόπο πρέπει να, να... να εφαρμόζεται το άρθρο 5 της συνθήκης της Ουάσιγκτον. Όπω γνωρίζετε υπήρξαν πάρα πολλέ συζητήσει για το άρθρο 5 που έχει δύο σημαντικέ αδυναμίες. Πρώτον, δεν εξασφαλίζει ότι οι δράσεις για την υποστήριξη ε, ενός ε, ε, κράτους που δέχεται επίθεση είναι ανεφόρον και θα σα πω και το εξή πάλι παράθεση από το άρθρο 5 λέει διάφορα μεταξύ των οποίων πρέπει να αποκαταστήσει την ασφάλεια της βορειοατλαντική περιοχής όχι όμως στην πρώτερη κατάσταση, στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την επίθεση σε ένα από τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ενδεχομένως η καλύτερη απάντηση να επιμείνουμε στην εφαρμογή του άρθρου 5 και η απάντηση πρέπει να είναι ανεφόρον, δεύτερον πρέπει να συνεχίσει μέχρι η κατάσταση, η πρώτερη κατάσταση πριν από την επίθεση αποκατασταθεί. Είναι ο μοναδικός τρόπος ε, με τον οποίο πρέπει να απαντήσουμε. Αυτό είναι ο σωστός τρόπος και αυτό είναι ένα ερώτημα προς τον κύριο Σία ε, καταρχάς. Να επανέλθω στη λεκάνη του ευξήνου πόντου. Δεν έχουμε μία πραγματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ για τον εύξηνο πόντο. Δεν έχουμε νέες στρατηγικές, δεν έχουμε πρόγραμμα. Απλώς αντιδρούμε σε αυτό που κάνει η Ρωσία. Απλώς αντιδρούμε. Σαν πυροσβέστες. Πρέπει να έχουμε μια μακροχρόνια στρατηγική για την περιοχή αυτή για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις ε, της κοινή ασφάλειας και άμυνας ε, και σε όλες τις απειλές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μίκα. Κύριε Κόλβιν Μίκα, έχω ένα ερώτημα προς τον κύριο Αστεβίτσιους είπε ότι η Ρωσία αποσταθεροποιεί την κατάσταση συγγνώμη, είναι ανταλλαγή απόψεων ε, μεταξύ των συναδέλφων ε, και των προσκεκλημένων μας. Μα είναι ένα πάρα πολύ σύντομο ερώτημα. Ε, λέτε ότι αποσταθεροποιεί την κατάσταση η Ρωσία και μετά λέτε εσείς ότι είναι αποσταθεροποιημένη ήδη η κατάσταση. Δεν κατάλαβα. Τι είναι καλό, η σταθεροποίηση τελικά ή η αποσταθεροποίηση. Δεν κατάλαβα ακριβώς αυτά που είπε. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ δεν έχει ζητηθεί ο λόγος από κανέναν άλλο συνάδελφο, οπότε θα ήθελα και εγώ να θέσω κάποια ερωτήματα. Καταρχάς, ε, ε, στον πρέσβη Ζανιέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι χρειάζεται προκειμένου να ε, ενισχύσουμε την αποστολή του ΟΗΕ του ΟΑΣΕ ε, υπάρχουν αποστολές παρατήρησης της κατάστασης ε, αποτελεσματικά. Παρακαλούμε να μας πείτε λίγα περισσότερα σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε και το σχόλιο μου προς τον κύριο Σέα. Προσφάτως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τη πολύ σημαντική έκθεση Λαντσπέργης για τη Ρωσία και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας όλοι οι σκιώδεις εισηγητές ε, συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό και ο ίδιος ο εισηγητής ε, προσπάθησαν να μην υπάρχει μνήα στην Ευρασιατική ε, Ένωση και την ενίσχυση της δικής μας εκτίμησης για αυτήν την ιδέα αναφέρεται μια ανοιχτή εναρμόνιση μεταξύ της Ένωσης και της Ευρωασιατικής Ευρασιατικής Ένωσης. μπορεί να αποτελεί απλώς μία παρεξήγηση ε, για τον ε, γενικό ε, γραμματέα, τον κύριο Σία. Θα ήθελα να πω επίσης ότι Εκτιμώ όλο ιδιαίτερο την προσέγγιση του ΝΑΤΟ για την αύξηση της ανθεκτικότητας ε, των τριών ε, κρατών, ε, Ουκρανία, Μολδαβία και Γεωργία, κατά του υβριδικού πολέμου που αποτελεί την ε, πολιτική αυτή τη στιγμή της Ρωσίας. Σίγουρα αυτές οι χώρες είναι πιο ευάλωτες από εμάς. Εμείς είμαστε εντός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και του ΝΑΤΟ. Τι μέσα θα μας συμβουλεύονται να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να αυξήσουμε αυτήν την αντοχή των χωρών αυτών. Υπάρχουν κάποια επιπρόσθετα ευρωπαϊκά μέσα εκτός από αυτά του ΝΑΤΟ τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατά την προσπάθειά μας αυτή. Δεύτερο ερώτημα, μια γενική παρατήρηση μάλλον για τις ε, παγωμένες συγκρούσεις. Για μένα είναι νέο το ότι ε, η αυτοανακηρυχθήσα κυβέρνηση, όπως αποκαλούμενη, ε, της περιοχής του Ντονιέσκ είναι ένας εμπειρογνώμονας πλέον, αυτό εγώ δεν το ήξερα και πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο να το γνωρίσει κανείς. Νομίζω ότι η ανταλλαγή πληροφοριών ε, των πληροφοριών που λαμβάνει το ε, ΝΑΤΟ για την παρουσία της Ρωσίας μπορεί να είναι πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί στην κοινοβουλευτική συνέλευση ε, του ΝΑΤΟ και η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κοινοβουλευτική αυτή συνέλευση μπορέσαμε να διαμορφώσουμε μία άποψη σχετικό σκηνή αρκετά προσφάτως και ακούσαμε και περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με την παρουσία της Ρωσίας στην Ουκρανία και μπορέσαμε να είχαμε περισσότερες πληροφορίες από αυτές που είναι διαθέσιμες ε, σε, σε άλλους φορείς. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους ανταλλαγή πληροφοριών που συνεισφέρει στις γνώσεις μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας δώσω τώρα το λόγο για να απαντήσετε. Κύριε Ζανιέ, έχετε το λόγο πρώτος. Ε, ευχαριστώ να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις του κυρίου Πρέντα για τις ε, συμφωνίες Μίνσκ και το θέμα το οποίο που έθεσε ο ε, συνάδελφος προσκεκλημένος. Δεν συμφωνώ απολύτως ε, με αυτό που είπατε ότι το Μίνσκ, οι συμφωνίες Μίνσκ οδηγούν σε, στις παγωμένες συγκρούσεις. Ε, εξαρτάται από το πώς εφαρμόζεται. Αν δούμε ε, τις ε, συζητήσεις, ε, συμφωνίες που έτυχαν διαπραγμάτευσης και άμα δει για παράδειγμα τις εκλογές που έγιναν στο πλαίσιο στις εκλογές και την εκλογική διαδικασία στην Ουκρανία και τις οποίες θεωρείται ότι ένας facilitator θα μπορούσε να τις παρακολουθεί ε, είναι διαφορετικό αυτό το ζήτημα ε, των εκλογών στις συγκεκριμένες περιοχές από τις εκλογές σε ολόκληρη την ε, Ουκρανία. Ίσως θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την εστίαση μόνο στην γραμμή ε, ε, ε, επαφών. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία από τις παγωμένες συγκρούσεις για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις δύο πλευρές και να δημιουργηθεί μια περιοχή η οποία θα έχει πλήρη αυτονομία αλλά θα αποτελεί τμήμα της Ουκρανίας και θα είναι κάτι για το οποίο όντως ναι, θα μπορούσαμε να διευκολύνουμε, κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να διευκολύνουμε ως παρατηρητές. Αλλά τότε το θέμα των συνόρων αφήνεται κατά μέρο για το τέλος και είναι σημαντικό για μα να μεταβούμε, να, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο το συντομότερο δυνατόν. Ε, το θέμα υπερβαίνει το ε, Μίνσκ ε, προσπαθούμε να βρούμε περιοχές ε, στις οποίες ε, η εκεχηρία δεν εφαρμόζεται για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε και υπάρχουν και πολλές, ε, υπάρχουν πολλοί τρόποι, απαντώ ε, σε ερώτηση που μου έγινε, ε, αλλά ένα σημείο αφεπηρίας είναι μερικές φορές μια στρεβλή θεώρηση που έχει ο ΟΑΣΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ΟΑΣΕ. Θεωρεί ότι είναι ένας εταίρος ο ΟΑΣΕ, αλλά πρέπει να δούμε τα πράγματα και από μια διαφορετική οπτική γωνία είναι μια πολύ σημαντική, ένας πολύ σημαντικός παίκτη εντός του ΟΑΣΕ. Είναι μια πλατφόρμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις δικές της πολιτικές, για τους δικούς της στόχους, όπως και η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το κάνουν όπου μπορούν. Ε, και μερικές φορές ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας ρωτά ε, πώς μπορούμε να έχουμε κοινέ πρωτοβουλίες ε, και ε, εμεί σας λέμε εσείς τι μπορείτε να κάνετε χρησιμοποιώντας τον ΟΑΣΕ. Έχουμε πάρα πολλές πρωτοβουλίες, πάρα πολλά μέσα, έχουμε τις ημέρες ασφαλείας, στις οποίες συμμετέχουν και οι εταίροι μας από τη Μεσόγειο, ε, πολιτισμικός διάλογος, ε, μπορούμε να ε, επεκτείνουμε κάπως την ημερήσια διάταξη αλλά και τους συμμετέχοντες, στους ξένους μαχητές για παράδειγμα ή την ριζοσπαστικοποίηση στην Κεντρική Ασία. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε. Μπορεί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στον ΟΑΣΕ αλλά να προσπαθεί να επιτύχει και τους δικούς της στόχους. Πρέπει να βλέπουμε κάπως ευρύτερα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας όπως έκανε ήταν για παράδειγμα στην Ουκρανία. Στην, η Ευρωπαϊκή Ένωση μα υποστήριξε πάρα πολύ στην εφαρμογή των πολιτικών μας, επιτόπου, ε, παρακολούθηση, ε, χρηματοδότηση που προήλθε σε μεγάλο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τώρα, όσον αφορά την απελευθέρωση των θεωρήσεων, κοιτάξτε, ε, αυτό αφορά και τις ε, ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Έχουν σημαντικό αντίκτυπο όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μέσα τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να μειώσουμε τον αντίκτυπο των συγκρούσεων. Το άνοιγμα των συνόρων είναι ένας τρόπος ενίσχυσης της σταθερότητας. Οπότε βεβαίως υπάρχει πάντοτε μία τεχνική πτυχή, αλλά δεν πρέπει να ε, εκλαμβάνεται μόνο ως τέτοια και ο πολιτικός αντίκτυπος είναι πάρα πολύ σημαντικός και γι' αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας και να το χρησιμοποιούμε για, ως εργαλείο. Η υπερδυνιστερία είναι ένα παράδειγμα ακριβώς αυτού του πράγματος οι σχέσεις ε, της οικονομικής δομής της υπερδνηστερίας με την Ευρώπη και με την, με, την υπόλοιπη Ευρώπη είναι επίσης πολύ σημαντικές. Και αν στο τέλος του έτους δούμε μια κατάσταση στην οποία θα χάσει το πλεονέκτημα του προνομιακού ε, εμπορίου ε, η υπερδνηστερία με την Ένωση, τότε θα δούμε ότι κάποιε εταιρείε, α πούμε μπορεί να καταχωρούνται στην Μολδαβία. Εμεί μπορούμε να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε ε, κατά αυτόν τον τρόπο ε, την επίλυση τη σύγκρουση. Ε, το ένα ερώτημα που μου έθεσε άλλο συνάδελφο αφορούσε τη Ρωσία και το οποίο το έθεσαν και άλλοι συνάδελφοι, όταν πρόκειται για τη σχέση τη Ρωσία με του γείτονε τη. Το ένα ζήτημα είναι ο τρόπο με τον οποίο βλέπει το θέμα η Ρωσία και το άλλο θέμα είναι πώ του βλέπουν οι γείτονε τους Ρώσους. Όπως γνωρίζετε, ε, οι περισσότεροι είναι και μέλη της ΟΑΣΕ. Εγώ είχα πάει στη Λευκορωσία, στο Καζακστάν, ε, ε, γνώρισα τον Υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας, είχα πάει πάρα πολλές φορές, ήμουν στην περιοχή σχεδόν συνέχεια κατά την περίοδο της κρίσης. Όμως, τελικά ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνει τις σχέσεις του με τη Ρωσία και αυτό το λέω σε σχέση και με το ερώτημα της αποστολής των αποστολών και ΕΠΑ ε, που μου ετέθη δεν είναι μόνο θέμα ενωσιακής πολιτικής αλλά και των χωρών αποδεκτών υπάρχει πάντοτε ένα κόστος σε κάθε απόφαση εξωτερικής πολιτικής. Αν μια χώρα θέλει να επενδύσει όλες τις σχέσεις της ε, προς μια κατεύθυνση, πάντοτε υπάρχει ένα κόστος σε σχέση με την έλλειψη σχέσεων ε, με, με κάπου αλλού. Ε, είναι μια απόφαση την οποία κάθε χώρα την παίρνει μόνη τη. Κάθε χώρα μπορεί να αποφασίσει πόσο θέλει να επενδύσει στη σχέση τη με τη Ρωσία εν προκειμένου ή με άλλου εταίρου. Και βλέπω ότι οι περισσότερες χώρες που γυπνιάζουν με τη Ρωσία ενδιαφέρονται στη διαφοροποίηση των σχέσεών του, αλλά με τρόπο ε, που μπορεί να αφορά οικονομικά συμφέροντα, συμφέροντα ασφαλείας, ε, πολιτική καλής γειτονίας. Θέλουν συχνά να διατηρήσουν μια καλή σχέση με τη Ρωσία, αλλά παρά αλλά θέλουν και να διαφοροποιήσουν και συν το χρόνο όλο και περισσότερο να βελτιώσουν τη σχέση τους ε, με άλλες χώρες. Και αυτό προσπαθείτε, πρέπει να μπείτε στη θέση αυτών των ανθρώπων για να μπορείτε να καταλάβετε ποιες είναι οι ενδιαφέρουσες χώρες προκειμένου να επενδύσετε, να προσπαθήσετε να επενδύσετε τη σχέση σας εννοώ, αλλά να προσπαθήσετε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργήσετε αποσταθεροποίηση. Και το λέω αυτό σε σχέση με την ιδέα της Γιάλτας που αναφέρθηκε προηγουμένως. Η Γιάλτα είναι ο κίνδυνος που βλέπουμε και προσπαθούμε φυσικά να καταπολεμήσουμε τον ε, κίνδυνο αυτό, γιατί διαφορετικά πάμε στη λογική του άρθρου 5 και ε, βεβαίως ε, έχουμε πολύ πιο προβληματικά σενάρια να αντιμετωπίσουμε το ερώτημα τώρα της ελευθερίας ε, ε κυκλοφορίας και επενδύσεων για τον ε, χιλίων ατόμων, των χιλίων ατόμων επιτόπου. Εμείς τώρα πηγαίνουμε προς τους 600. Ελπίζω να φτάσουμε τους 600 κάτι διάρκεια του καλοκαιριού. Ο αριθμός θα παραμείνει σε σχέση βέβαια με το τι μπορούμε να κάνουμε ε, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιτόπου αν δεν υπάρχει το περιθώριο να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Χρειαζόμαστε δηλαδή μεγαλύτερη ελευθερία κυκλοφορίας και πρόσβαση στο σύνορο. Δεν έχουμε πρόσβαση στα σύνορα αυτή τη στιγμή γιατί οι αυτονομιστές μας ε, ε, μπλοκάρουν. Οι Ρώσοι μας λένε εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, συζητήστε εσείς με τους αυτονομιστές, εκείνοι είναι που αποφασίζουν. Ε, και επομένως εμάς μας μπλοκάρουν. Έχουμε, παρακολου... Έχουμε ανθρώπους που παρακολουθούν οι οποίοι είναι άμαχοι, ε, δεν έχουν όπλα και αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα σε τάγκς και με όπλα που προσπαθούν να μας, ε, προσπαθούν να μας... δεν μας αφήνουν να περάσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Ούτε μπορώ εγώ να διακινδυνεύσω να μας πάρουν όμοιρους ε, ε, άνθρωποι με όπλα και τάγκς. Ε, και η Ρωσία έχει αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Επομένως, έχουμε ένα σχέδιο σιγά σιγά να απομακρύνουμε τον κόσμο, αλλά πρέπει να δούμε και τις συνθήκες επιτόπου που να το δικαιολογούν, γιατί είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με το θέμα της ασφάλειας. Δεν θέλουμε οι παρατηρητές μας να ε, τεθούν σε κίνδυνο. Μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να μην υπάρξουν ε, ε, σοβαρά προβλήματα. 70% των παρατηρητών προέρχονται από χώρες της Ένωσης και φυσικά πρέπει να τους φροντίσουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Το σχέδιο αύξησης υπάρχει αλλά δεν θα γίνει εν μία ανοιχτή. Η παρουσία τώρα των Ρώσων. Έχουμε μία αποστολή περίπου 500 παρατηρητών και 20 Ρώσοι ε, μεταξύ των 500. Δεν είναι μία ομάδα Ρώ, δεν, υπά... δεν υπάρχουν ομάδες Ρώσων, αλλά που και που εμφανίζεται και ένας Ρώσος, ε, συνήθως είναι τέσσερις παρατηρητές ε, ε, μπορεί να είναι ένας Ρώσος, ένας Αμερικανός, ένας Νορβηγός και ένας Ιταλός που επιβαίνουν στο ίδιο αυτοκίνητο, ένας οδηγεί και οι άλλοι κάθονται. Όταν όμως βρίσκομαι σε περιοχές ε, αποσχιστικές, ε, ε, μερικές φορές είναι σημαντικό να έχουμε Ρώσους γιατί έτσι έχουμε καλύτερη επαφή, μπορούμε καλύτερα να ε, συζητήσουμε με κάποιους ε, από τους Ρώσους μαχητές ή με τον τοπικό πληθυσμό. Και αυτό δεν είναι κακό από απόψεως αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Προσπαθούμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε συγκέντρωση συγκεκριμένων ε, εθνικών ομάδων κάπου. Έχουμε Ρώσους όχι μόνο στην Ατολή αλλά και σε άλλες περιοχές. Και αυτό είναι αυτό που κάνουμε ε, στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ, είναι ότι αν δεν έχουμε αυτήν την κατανομή στις εθνικότητες, μετά είναι σαν να γινόμαστε ΝΑΤΟ. Εμείς προσπαθούμε να υπάρχει μια συνένεση και όλοι να συμφωνούν με όλα αυτά που κάνουμε. Αυτό είναι η φύση των όσων προσπαθούμε να κάνουμε. Αν δεν θέλετε κάποιες χώρες να μπουν σε μια επιχείρηση τέτοιου είδους, ε, τότε δεν χρειάζεστε τον ΟΑΣΕ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΟΑΣΕ αυτό το πλαίσιο έχει και ε, προσπαθούμε και από αριθμητική απόψεως να διατηρήσουμε αυτήν την ισορροπία και προσπαθούμε να είμαστε και αντικειμενικοί στην έκθεση. Όλοι συμφωνούν στην υποβολή εκθέσεων, ε, δεν ε, αφορά μια συγκεκριμένη εθνικότητα, λαμβάνουμε υπόψη όλα όσα μας λένε. I think this... Νομίζω ότι αυτό καλύπτει την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας ε, το λαμβάνω υπόψη μου, αλλά είναι ένας τομέας όπου μέσω των παγωμένων σειράξεων ε, συνεχίζουμε να προσδίδουμε μεγάλη σημασία σε αυτή την περιοχή. Ευχαριστούμε τον πρέσβη. Ε, ο Γενικός Γραμματέας έχει το λόγο. Όπως ξέρετε, στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο κάνουμε ενημερώσεις και πολλές φορές ανακύπτουν γύρω στις 25-30 ερωτήσεις. Και το δύσκολο είναι να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις χωρίς να τα ταπανίσουμε πολύ χρόνο. Ο Λαμπέρτο ευτυχώς απάντησε αρκετές και με τον, ε, μπορώ να αφήσω τα ε, υπόλοιπα στον James, τον κύριο Σερ. CSR, ε, υπάρχει σύγχυση με τα ονόματά μας. σε σχέση με το θέμα της Ρωσίας, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά ψευδοσχήματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ρωσία εξάγει 60, 160 δις κυβικά μέτρα. Και γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν μπορεί η Κίνα να υποκαταστήσει αυτή την αγορά και ίσως οι δύο πλατφόρμες που έπρεπε να χτιστούν, να μην χτιστούν, γιατί υπάρχει σχιστολιθικό αέριο στην Κίνα, απομακρύνει τον άνθρακα από την οικονομία της, παράγει και ηλιακή ενέργεια και σίγουρα από το υγροποιημένο φυσικό αέριο έχει μια αγορά. Αλλά η Ρωσία πιστεύει ότι υπάρχει μέλλον στους υδρογονάνθρακες στην Ασία γιατί μειώνεται η αγορά στην Ευρώπη λόγω ανανεώσιμων και η Κίνα προβάλλει τις ανανεώσιμες γι' αυτό θα ε, καθυστερήσει η οικονομία για 20-30 χρόνια. Γι' αυτό η Ρωσία θα ακολουθήσει πτωτική τάση. Ε, θα έχει, δεν θα έχει την ίδια δύναμη μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, διότι οι υδρογονάνθρακες ε, δεν έχουν το, το ίδιο μέλλον και σίγουρα η Ρωσία θα είναι εταίρος της Κίνας, αλλά σε χαμηλότερη κλίμακα. Σε σχέση με τις χώρες BRICS, μπορώ να πω ότι στην ΟΥΦΟ, στην ε, ε, διάσκεψη της προηγούμενης εβδομάδας, είδαμε ότι η Ινδία και το Πακιστάν χτυπάν την πόρτα και βλέπουμε ότι επεκτείνεται ολοένα και η Νότιος Αφρική. Ποιος ξέρει, ίσως και το Ιράν αύριο. Άρα η ρωσική επιρροή μειώνεται και θεωρώ ότι η επιρροή της Κίνας θα αυξηθεί. Η ε, Τράπεζα Ανάπτυξης των BRICS και αυτή η νέα αναπτυξιακή τράπεζα της Κίνας δείχνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πλατφόρμες όταν μιλήσουμε με την Ινδία, το Πακιστάν, τις χώρες BRICS, τη στιγμή που θέλουμε να φτάσουμε σε άλλα φόρα τα οποία είναι πιο δελεαστικά. Δηλαδή το BRICS, τα BRICS δεν είναι μία συνεκτική οντότητα. Αποτελούν το 20% ε, output πετρελαίου, αλλά ε, το πρόβλημα του πετρελαίου για τη Ρωσία παραμένει. Γι' αυτό θα μπορούσα να πω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε, να προωθήσουμε το TTIP, γιατί θα φέρει ανάπτυξη και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Και μετά υπό επιφυλάξεις. Ε, χαίρομαι διότι το Κογκρέσο οδήγησε σε μια διαδικασία fast track την προηγούμενη εβδομάδα για ένα TTIP με την Ασία. Θα πρέπει να προωθήσουμε αυτές τις συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων. Και δεν νομίζω ότι η Ασία είναι υποκατάστατο ε, στην ηγεμονία της Ρωσίας και δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολύ ε, πολλές ολιγαρχικές ομάδες εκεί. Τρία εκατομμύρια Ρώσοι έφυγαν από τη Ρωσία. Οι περισσότεροι εργάζονται στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ. Άρθρο 5. Αυτοματοποιημένο σύστημα. Δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Και θα σας πει. Φανταστείτε τη χώρα σας, ας πούμε μια χώρα του ΝΑΤΟ. Ξαφνικά Τη τηλεφωνεί άλλος σύμμαχος που λέει έχω τι επίθεση στον κυβερνοχώρο, έχει πέσει το ηλεκτρικό μου δίκτυο και θέλω αύριο να εκινήσω την ε, διαδικασία του άρθρου 5. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί ένας ε, σύμμαχος να οδηγήσει, στην, να οδηγήσει ένα άλλο σύμμαχο να συμμετέχει σε μία διαδικασία του άρθρου 5. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει αυτό όταν πρόκειται για δύο χώρες της ε, ίδιας συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, ε, δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο να ξεκινήσει ε, μία διαδικασία πολέμου επειδή το κρίνει ένας σύμμαχος και να συμπαρασύρει και έναν άλλο. Διότι το άρθρο 5 το επικαλούμαστε μόνο εκεί που αιτιολογείται. Αλλά στην περίπτωση του Κωσυφοπεδίου, Αφγανιστάν, Λιβύη στην αρχή το ΝΑΤΟ έδρασε πάντα σωστά. Μετά την 11η ε, Σεπτεμβρίου έδρασε σωστά το ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο η αξιοπιστία μας είναι σωστή. Αν δεν υπάρχει αλληλεγγύη δεν θα φτάσουμε εκεί. Γιατί πιστεύετε ότι αυτά τα στρατιωτικά σχέδια και ασχέδια ασκήσεις ε, προωθήθηκαν σε σχέση με την θέση των εξοπλισμών. Τώρα θα έχουμε ένα νέο στρατηγείο του ΝΑΤΟ σε όλα τα κράτη-μέλη, σε όλα τα κράτη. Ε, άμεσες απαντήσεις, ε, άμεση προειδοποίηση. Γιατί ετοιμαζόμαστε για την μεγάλη στιγμή. Έχουμε εξοπλισμό, υποδομή, στρατιωτικές δυνάμεις. Ο καθένας ξέρει το ρόλο του τη σωστή στιγμή. Και όταν κάνετε ασκήσεις έστω επί χάρτου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την κατάσταση τη σωστή στιγμή. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ε, την αιρεσιμότητα έτσι όπως τη θεωρούσαμε. Ως προς την ε, ε, μαύρη θάλασσα για τη Βαλτική ήταν ήσυχες περιοχές, τόσο ήσυχες που δεν προωθήσαμε τις θαλάσσιες ικανότητές μας εκεί. Τώρα ε, έχουμε έλλειψη ε, πλοίων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η Royal Navy είχε ε, γύρω στα 373. Τώρα έχουμε 18-19 λειτουργικά πλοία, πολεμικά πλοία. Δεν μιλάμε για το Mare Nostrum με τον ίδιο τρόπο, γιατί στην Ανατολική Μεσόγειο η Ρωσία ελέγχει περισσότερο την ακτογραμμή της ε, Κασπίας θάλασσας και της ε, Μαύρης θάλασσας. Αυτό αφορά και την εγκατάσταση, τις εγκαταστάσεις στην Κρυμαία και στο Καλίνιγκραντ έτσι ώστε να μπορέσει η Ρωσία να ελέγχει το παιχνίδι σε αυτά τα απομακρυσμένα σημεία ως προς τις πυραυλικές εγκαταστάσεις. Και υπάρχει και το Anti-Access Aerial Denial Υπάρχουν σύμμαχοι η Γεωργία, η Ουκρανία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία στην Μαύρη Θάλασσα και θα πρέπει να έχουμε ε, πρόσβαση. Πρόκειται για ένα μεγάλο στρατηγικό θέατρο. Τώρα κατά πόσο χρειαζόμαστε μια θαλάσσια στρατηγική, μια στρατηγική της Μαύρης Θάλασσας, αυτό είναι ένα διαφορετικό ζήτημα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια περιπολία ως προς το θέμα της ε, ανθεκτικότητας είδαμε το θέμα των, ε, της συμμετοχής των διαφόρων κέντρων και μονάδων ιδιαίτερα ως προς τα ηλεκτρικά δίκτυα. Μιλάμε για την ασφάλεια των δικτύων, ιδιαίτερα από πλευράς ε, Ουκρανίας. Δυστυχώς δεν υπάρχει ασφάλεια. Υπάρχει μια συνεχής διείσδυση. η Ρωσία γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση της Ουκρανίας και τώρα με την επιμελητιακή βοήθεια ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Εστιάζουμε την προσοχή μας στη δική μας ανθεκτικότητα και ελπίζουμε να βοηθήσουμε και τους συμμάχους. Ως προς τις παγωμένες ε, σειράξεις, δεν είναι παγωμένες οι σειράξεις, αλλά οι διαπραγματεύσεις. Και στον Αγκόρνο ε, ε, Καραμπάχ είχαμε 60 νεκρούς πέρσι από ελεύθερους σκοπευτές και το είδαμε και στην πρώην Ιουκοσλαβία. Είδαμε τι έγινε το 1995, μπορούν να ξαναανοίξουν ε, οι σειράξεις. Γι' αυτό η παρουσία είναι ζωτικής ε, σημασίας, κίνητρα και κυρώσεις έτσι ώστε οι σύμμαχοι να επιλύουν τις σειράξεις και να επαγρυπνούμε διότι επικεντρωνόμαστε σε μία κρίση που, που ξεχνάμε μία γειτονική κρίση και στην Ευρώπη θα πρέπει να είμαστε πολυεπίπεδοι, δηλαδή να εχουμε τεσσερα τέσσερα-πέντε προγράμματα όπως την τηλεόραση και να τα παρακολουθούμε παράλληλα. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου 4 ή 5 καταστάσεις, αλλά τη στιγμή που έχουμε ένα προετοιμασμένο μέτρο θα τα καταφέρουμε. Η Μαριούπολη τώρα. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι ετοίμασε ένα πακέτο νέων κυρώσεων και είναι σίγουρο το τι θα συμβεί αν υπάρξει κλιμάκωση. Οποιοςδήποτε ε, επιτιθέμενος θα πρέπει να κάνει αυτή την αποτίμηση κόστους ωφελίας. Και στην περίπτωση της Μαριούπολης θα έχουμε κλιμάκωση που σημαίνει ότι η Ρωσία δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό κρυφά και θα πρέπει να επιβαρυνθεί με τις επιπτώσεις. Ας ελπίσουμε ότι το οικονομικό πακέτο θα είναι αρκετά αναχαιτιστικό και σταθεροποιητικό. Αλλά από την κατάσταση ένα χρόνο πριν ε, καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε και για τα χειρότερα δυνατά σενάρια. Thank you, sir. Mr. Scher. Thank you, Madam Chairman. Let me start with ο κ. Σέρ. Πρώτα, δύο διαπιστώσεις, ένα τρίτο για το Μίνσκ και να επανέλθω σε τρεις γενικότερες ερωτήσεις. Πρώτο, δεν είχα την πρόθεση να πω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε επίσημες συνομιλίες με την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση. Δεν είπα αυτό. Υπάρχουν όμως ειδήσει από ποιοτικά έγγραφα του διεθνούς τύπου που λένε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμέρους Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δεσμευτεί καταρχήν να προχωρήσουν σε κάποιο είδους συνομιλίες για εναρμόνιση και για αντιμετώπιση των διαφορών μας με την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση. Για το στρατηγό Αντουφίβ. Αυτός διορίστηκε το 2014 όταν οι αποσχιστές ητώνταν. Δεν γνωρίζω αν ακόμα κατέχει τη θέση του και νομίζω ότι είναι αδύνατο να το μάθει κανείς. Για τους άλλους που λειτουργούν εκεί δεν έχουν την ίδια τεχνογνωσία. Υπάρχουν βέβαια ρωσικέ ειδικέ δυνάμεις που έχουν σχετική τεχνογνωσία. Ο κύριος Κίρκιν, Συνταγματάρχη, που ήταν και παλαιά υπουργό Άμυνα, έχει μακρά εμπειρία από αγώνες στην Τσετσενία και ούτε καθεξής. Τα έχει μέσα στο DNA του λοιπόν. Τώρα, το Μίνσκ λέει καθαρά, η συμφωνία Μίνσκ δηλαδή, ότι οι αποφάσεις όχι μόνο για την ανάκτηση του ελέγχου των συνόρων της Ουκρανίας, αλλά και οι διατάξεις σχετικές με, την, με τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και τις εκλογές. Πρέπει να συμφωνηθούν με τις τοπικές αρχές. Το κείμενο στα ρωσικά λέει κάτι που είναι κάπου μεταξύ διαβούλευσης και συντονισμού. Επίσης δεν αναφέρεται σε αποκέντρωση, αλλά στην καθίδρυση καθεστώτων, ειδικών καθεστώτων στις περιοχές αυτές. Και σε αυτό αναφερόμουν πριν. Τώρα, ας συνοψίσω ορισμένες σχετικές ερωτήσεις. Κύριε Γκάλερ, πρώτον, είπατε ότι η Ρωσία δεν διαθέτει ελκυστικότητα. να αμφισβητήσω λίγο αυτό που λέτε και να με συμπαθάτε. Ίσως να μην έχει ελκυστικότητα το ρωσικό κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο. Όμως πολιτικά η Ρωσία διαθέτει ελκυστικότητα. Διότι έχει εμφανιστεί ως ο σημεοφόρος όλων εκείνων στην Ευρώπη αλλά και αλλού που αντιτίθεται σε αυτά που αποκαλεί ο Λαυρόφ δυτικός μεσιανισμός. Αντιτίθεται σε, αυτό τον φιλελεύθερο, σε αυτή τη φιλελεύθερη συνένεση στην Ευρώπη. Και σε αυτά έχουν επενδύσει, επανέρχομαι σε αυτό που είπε ο Τάνοκ. Σε μία, να εμφανιστούν δηλαδή ως μία δύναμη αντι-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί πολλοί βρίσκουν τη ρωσική στήριξη πολύ ελκυστική. Δεύτερο, τι εννοούσα όταν είπα να προετοιμαστείτε για εκπλήξεις. Δεν έχω κρυμμένο τίποτα στο μανίκι μου, θα σας εξηγήσω γιατί το είπα. Πρώτο, δεν μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα εδώ βέβαια πλήρως. Υπάρχουν κάποιες τάσεις και κάποιες εντάσεις μέσα στο ρωσικό στρατιωτικό σύστημα που τους προκαλεί προβλήματα. Υπάρχει μεγαλύτερο εξαναγκασμός μέσα στο ρωσικό στρατιωτικό σύστημα για να τους κρατήσουν επί τόπου αυτούς που τους στέλνουν. Και υπάρχει και μικρή έκθεση εθνικών ρωσικών στρατευμάτων σε εχθρικές, εχθρικά διακείμενες δηλαδή τοπικές κοινωνίες. Και ως αποτέλεσμα υπάρχει μία, ένας δισταγμός να αναμειχθούν σε μακροπρόθεσμες πολεμικές σειράξεις. Αυτό που έχουν μάθει να κάνουν είναι να παρεμβαίνουν, να επεμβαίνουν με δυναμικό τρόπο να καταστρέφουν την, ε, τις αντιτιθέμενες δυνάμεις και να αποχωρούν. Αυτό κάνει οι ρωσικές δυνάμεις. Αυτό που γίνεται τώρα νομίζω είναι ότι κάθεται και σκέπτονται ποια να είναι η επόμενη κίνησή τους όχι αν θα διατηρήσουν το status quo και θα το δεχτούν. Γίνεται μια αξιολόγηση, αυτό που λένε οι Αμερικανοί, ότι όλες οι επιλογές είναι επιτάπητος για το Κρεμλίνο. Λέγουν και προλέγουν ότι δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην Ουκρανία, διότι λένε η Ουκρανία είναι τεχνητό κράτος, δεν έχει πραγματικά θεμέλια, αλλά διατηρείται η σταθεροποίηση. Αυτοί θεωρούν ότι αν του δώσουν άλλη μια σκοπιά θα καταρρεύσει το σύνολο του οικοδομήματος και όμως δεν καταρρεύει. Ίσως λοιπόν να επιμείνουν περισσότερο, ίσως να προχωρήσουν σε άλλες πολεμικές δράσεις, να χρησιμοποιήσουν κάποιες δυνάμεις τους υπό άλλη ιδιότητα κάπου αλλού, μπορεί να ανταποκρίνονται ασυμμετρικά πολλές επιλογές τις οποίες μπορούν ενδεχομένως να υποστηρίζουν με κάποιες περιστασιακές ενδείξεις. Τι πάση δηλαδή κάποιων περιστασιακών ενδείξεων. Τέλος, γιατί βέβαια το ρολόι προχωρεί, για το θέμα της σταθεροποίησης. Είναι δυνατό να διατηρηθεί στρατιωτικό ε, status quo χωρίς την προμήθεια εξοπλισμών. Εγώ θεωρώ ότι οι κυρώσεις αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για να συγκρατήσουν τη συμπεριφορά των Ρώσων. Οι κυρώσεις αποτελούν πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την μείωση της ρωσικής ικανότητας, capacity, σε σημαντικούς τομείς και την μείωση της ικανότητας εξυγχρονισμού. Αυτό όμως που βλέπουμε από τις συμφωνίες Μίνσκ 1 και 2, μετά από την εντατικοποίηση δηλαδή των κυρώσεων, μετά από τις επιθέσεις, είναι ότι έως τώρα δεν έχουν περιορίσει, δεν έχουν συγκρατήσει την συμπεριφορά των Ρώσων. Χρειάζεται λοιπόν μια σοβαρή συζήτηση που διεξάγεται αλλού για το πώς να δημιουργηθεί μια δομή συγκράτησης και αποτροπής εντός της Ουκρανίας που θα περιλάβει ποικιλία μέτρων για την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας. Πολλά από αυτά γίνονται. Η Ουκρανία λαμβάνει και από διάφορες δυτικές χώρες αυξανόμενο αριθμό εξοπλισμών παρόλο που δεν τις βάζουμε στο, στην κατηγορία θανατηφόρων όπλων. Και ορισμένα από αυτά μπορούν να προκαλέσουν τη Ρωσία, θεώρησαν ορισμένοι. Ωστόσο, δεν το έχουν κάνει. Ο Πούτιν προκαλείται μόνο από μπλόφες και από ένδειξη αδυναμία. Αυτό είναι το τελευταίο. Λαμβάνει το μικρόφωνο κυρία Φωτίγκα, Προεδρεύουσα. Μία μικρή προσθήκη κυρία Πρόεδρε. Ίσως να μην σας αρέσει αυτό που θα πω τώρα. Γι' αυτό θεωρώ ότι εάν είχαμε δώσει υποστήριξη στην Γεωργία και στην Ουκρανία θα είχαμε το ίδιο, τα παλιότερα δηλαδή θα είχαμε δει τα ίδια γιατί η Ρωσία βλέπει ότι δεν έχει το ΝΑΤΟ την πολιτική βούληση για να προχωρήσει σε δράση. Το θεωρούν μπλόφα λοιπόν. Και αν δείτε το ιστορικό του Πούτιν, ποτέ δεν θα βρείτε να έχει χρησιμοποιήσει βία κατά ισχυρότερου αντιπάλου. Μάλιστα, σας ευχαριστώ αγαπητέ κύριε, λέει η κυρία Φωτίγκα. Ευχαριστώ και ιδιαίτερως για την τελευταία αυτή φράση που είπατε και να μου επιτρέψετε να την αναπτύξω λίγο προχωρώντας στην ε, συναγωγή των συμπερασμάτων και έχω να πω τρία πράγματα Πρώτο, η συμφωνία με το Ιράν, ανακοινώθηκε η συμφωνία με το Ιράν, μόλις τώρα, και θεωρώ, μάλλον διαρωτώ με ποιο θα είναι το τίμημα για την επικοδομητική στάση της Ρωσίας στην συμφωνία αυτή. Το πρόβλημα και ο κίνδυνος στη γενική εικόνα είναι που βλέπουμε τη Ρωσία τόσο επικοδομητική σε πολλά μέρη του κόσμου. Δεν αναφέραμε την Κρυμαία, ούτε μια φορά σήμερα. Όμως όλοι και όλες συμφωνούμε ότι πρόκειται για καθαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου η προσάρτησή της δηλαδή. Και πρόσφατα ένας από τους εταίρους μας χρησιμοποίησε καθαρή βία για να προσαρτήσει τμήμα της εδαφικής επικράτειας, επικράτειας γειτονική μας χώρας. Πρέπει λοιπόν να καθίσουμε να σκεφτούμε για ένα αποτελεσματικό οπλοστάσιο, η εργαλεία, η μέσα, για να αποτρέψουμε την Ρωσία και να φύγει από τη γειτονιά μας. Έχω ξαναπεί ότι εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω για τους υπόλοιπους. Εγώ, ωστόσο, η κατοικία μου είναι 200 χιλιόμετρα από τη ζώνη του Καλίνιγκρατ και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου δεν θεωρούμε ότι είναι ευχάριστο πράγμα αυτό. Δεν πιστεύω να το δούμε ποτέ αυτό στην Πολωνία, αλλά οφείλουμε να προβληματιστούμε σχετικά με αποτελεσματικά μέσα αποτροπής έναντι της Ρωσίας. Σίγουρα ήταν πολύ ενδιαφέρον που παρακολουθήσαμε την τοποθέτηση του πρέσβεως κ. Ζανιέ σχετικά με το τι σημαίνει το monitoring του ΟΑΣΕ είτε μας αρέσει είτε όχι πρόκειται για οργανισμό που συμπεριλαμβάνει πολλές χώρες, στην, οποίε συμμετέχει και η Ρωσία, που προχωρεί με συνένεση και πρέπει να σκεφτούμε αν θα προσφύγουμε και σε άλλα μέσα. Γιατί είμαι βεβαίω ότι η Ουκρανία φοβάται αυτή την ρωσική συνιστόσα μέσα στο monitoring. Τα ακούσαμε αυτά και στη διάρκεια των αποστολών που κάναμε στην Ουκρανία ως ε, η υποεπιτροπή. Άμυνας και ασφάλειας. Γνωρίζοντας και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η Ρωσία, σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ικανότητά, μας παρακολούθησης, monitoring δηλαδή, γιατί η παρουσία των Ρώσων παρατηρητών, έστω και αν ανέρχονται μόνο στο 1 τέταρτο, 1 πέμπτο. 1 πέμπτο λέτε, τη συνολική δυνάμεως. Α, 5% λέτε. Ωστόσο, εξακολουθούν να είναι ένα πρόβλημα, εφόσον προέρχονται από τον επιτιθέμενο. Ο επιτιθέμενος έρχεται και παρακολουθεί την ασφάλεια στο κατεχόμενο έδαφος. Αυτή είναι η εικόνα τελικά. Σας ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.